the speaker. Yeah. <laughs> Okay, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ και ευχαριστώ όλους όσους κατάφεραν να έρθουν παρά την απεργία, την ακύρωση των πτήσεων, τα προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, μερικοί έκαναν μεγάλο δρόμο για να καταφέρουν να έρθουν στη συνεδρίαση. Αλλά δεν μπορούσαμε να αναβάλουμε τη συνεδρίαση γιατί δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Σημείο πρώτο. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχει κατατεθεί πρόταση για το 9 της Εργασίας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Εκπροσώπησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης του κυρίου Σαρλ Γκέρανς έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ο ίδιος ο εισηγητής πρότεινε να αφαιρεθεί το σημείο αυτό την ημερήσια διάταξη θα το αφήσουμε για τη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, οπότε μπορούμε να βάλουμε αυτό το σημείο για άλλη φορά, για το Φεβρουάριο. Επίσης, δεν έχουμε βέβαια εκπροσώπους όλων των ομάδων, θα πρότεινα να αντικαταστήσουμε αυτό το σημείο με τα δύο τελευταία της εκθέσης Νόιζερ δηλαδή για την Συμφωνία σύμπραξης, αλληλευτική σύμπραξη με τη Σενεγάλη. Ο κύριος Νόιζερ συμφωνεί να συζητήσουμε νωρίτερα αυτά τα σημεία, ώστε να ψηφίσουμε και νωρίτερα, δηλαδή πριν έρθει ο Επίτροπος Μίμητσα. Ενημερώστε παρακαλώ τα μέλη. Μία ψηφοφορία, το θέμα δεν είναι επίμαχο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τις 6 και 4 μόνο και μόνο για να ψηφίσουμε. Παρακαλώ ενημερώστε εγκαίρως τα μέλη των ομάδων, ώστε να ψηφίσουμε 6 ε, και 4, ε, και 4. 4 και 4, 4,5 να ψηφίσουμε πριν τη συζήτηση με τον Επίτροπο Μίμητσα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να τελειώσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Μιμίτσα για να ψηφίσουμε. Οπότε, διαγράφουμε το 9, μετατοπίζουμε τα 11 και 12 πριν από το, την ανταλλαγή απόψεων με το Μίμητσα και με αυτές τις αλλαγές εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2, έγκριση των πρακτικών. Πρακτικά της 3ης Νοεμβρίου. Τα έχετε λάβει τις παρατηρήσεις στη γραμματεία πριν το τέλος συνεδρίασης. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, μέχρι το τέλος συνεδρίασης θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ανακοινώσει της Πρόεδρου. Την Πέμπτη το πρωί σε 9 θα γίνει κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού με θέμα την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ΑΕΤ. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Νέβεν Μίμητσα για την διαδικασία απαλλαγής. Έχουν προσκληθεί και τα μέλη της Επιτροπής μας. Η συνεδρίαση θα γίνει την 5η το πρωί σε 9, όπως σας είπα, στην αίθουσα 4Q1. Παρακαλώ, υπενθυμίστε στους συναδέλφους αυτή την συνάντηση. Θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την ΑΕΤ. Πολύ σημαντική συζήτηση στην αίθουσα 4Q1, 9 το πρωί της 5ης. Αυτή ήταν η μία και μοναδική ανακοίνωση που είχα. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5, ώρα των ερωτήσεων. Δεν έχουμε ανακοινώσεις της ε, Επιτροπής, γιατί θα έρθει ο ίδιος ο Επίτροπος ε, αργότερα στις 4.30. Ε, οπότε ανακοινώσεις Επιτροπής δεν έχουμε. Πάμε στο 5, ώρα των ερωτήσεων. Δεν έχουν κοινοποιηθεί ερωτήσεις. Άρα πάει και το 5 και περνάμε κάθε στο 6. Συζήτηση για την απαλλαγή του 2013 στον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρότεινα το θέμα του Γενικού Προϋπολογισμού και την απαλλαγή για το Αναπτυξιακό Ταμείο να τα συζητήσουμε μαζί για να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή της συζήτησης. Ε, ο προηγούμενος ηγητής ε, δεν επανεξελέγει, οπότε ανέλαβα εγώ ως πρόεδρος τις δύο αυτές εκθέσεις απαλλαγής. Να σταθώ σε λίγα σημεία των δύο εκθέσεων που έχετε λάβει για την απαλλαγή 2013 για το Γενικό Προϋπολογισμό και το Αναπτυξιακό Ταμείο. Καταρχήν, για το Γενικό Προϋπολογισμό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι για τη νέα εστίαση της Επιτροπής ε, ε, του προγράμματος σε, στις επιδόσεις. Γιατί παλιά απλώς ήταν μια ποσοτική ε, καταμέτρηση, τώρα γίνεται και ποιοτική αξιολόγηση του κατά πόσο πιάνουν τόπο τα χρήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βασικό πρόβλημα της ε, εκτέλεσης, όπως ξέρουμε, είναι η έλλειψη των πιστώσεων πληρωμών για πολλές δημοσιονομικές γραμμές που αφορούν ανθρωπιστική βοήθεια. Το συζητήσαμε και προηγουμένως με τον προηγούμενο Επίτροπο και η έλλειψη αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις Γενικές Διευθύνσεις ΔΕΦΚΟ και ΕΚΟ. Γιατί πάλι αφιερώνουν πολύ χρόνο στη μεταφορά κονδύλων από τη μία γραμμή στην άλλη και αυτή η δημοσιονομική διαχείριση αμαυρώνει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κανονικά είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης γίνονται οι περίμενες καθυστερημένες πληρωμές, παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Είναι κρίμα. Οπότε ελπίζω στο νέο προϋπολογισμό και το 2015 να καλυφθούν αυτά τα προβλήματα. Επίσης έχουμε τις αντιπροσωπίες. Σημαντικό θέμα. Και εδώ θα πρέπει η έλλειψη προσωπικού να αυξήσει το ποσοστό σφάλματος σε ό,τι αφορά τη χρήση της, ε, βοήθειας, της ευρωπιστικής βοήθειας και την δρομολόγησή της. Επίσης, απαλλαγή για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης. Ε, μείωση της φτώχειας καταρχήν στην υποσαχάριο Αφρική. Είναι θέμα και τη, των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Βέβαια, δεν είναι το αναπτυξιακό ταμείο μόνος το μόνο εργαλείο για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, αλλά σίγουρα συμβάλλει με αξιόπιστο τρόπο στην υλοποίηση. Έχουμε ένα σημαντικό νέο τρόπο για, τον, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας στις χώρες ΑΚΕ. επισημαίνει την πρόοδο και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε μια νέα προσέγγιση για τον προϋπολογισμό του 2013 και ελπίζω ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Δεμέλο, της ΔΕΦΚΟ, για να μας μιλήσει τον Ιανουάριο για τη δημοσιονομική στήριξη προς τις χώρες, ε, ε, πώς λειτουργεί, πώς το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης να απαντήσει σε απορίες ε, ή να διασκεδάσει αμφιβολίες των μελών για το θέμα της δημοσιονομικής στήριξης. Αυτά. Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Γκερέρο. Άλλος κανείς για να συντάξουμε κατάλογο μιλητών. Γκέρενς. Πρώτα Ερίκε. Ε. Ευχαριστώ Λίντα. Όχι μόνο για την παρουσίαση που μας έκανες μόλις, αλλά και για το γεγονός ότι ανέλαβες μια ευθύνη που σου αναλογεί ως πρόεδρος της Επιτροπής, γιατί ο προηγούμενος ηγετής απεχώρησε, δεν επανεξελέγει. Το θέμα τώρα για τη διαχείριση του προπολογισμού είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και θα το συζητήσουμε και με τον Επίτροπο, τον κύριο Μίμητσα, θα έχουμε την ευκαιρία. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα του Κοινοβουλίου και σε κάποιο βαθμό οδηγεί σε αποτελμάτωση ε, και αποτελεί τροχοπέδι για πολλές δραστηριότητες αυτή τη στιγμή έχει βλοκαριστεί ο προπολογισμό για το 2015 γιατί ακόμα δεν έχουν λυθεί οι εκκρεμεί πληρωμέ του 2014. Και κάθε χρόνο συζητάμε για ένα χρόνο ολόκληρο σχεδόν για θέματα ε, που έχουν ήδη εκτελεστεί και δεν έχουν ε, χρηματοδοτηθεί, δεν έχουν εξοφληθεί. Και μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο. Το έλλειμμα περνάει από το ένα έτος στο άλλο. Και ε, ουσιαστικά αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους ως Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά και γενικότερα τη χρηματοδότηση της Ένωσης, ε, ιδιαίτερα τις σχέσεις του Κοινοβουλίου με όλα αυτά. Διότι είναι συνομοθέτης για τον προπολογισμό. Συγκεκριμένα τώρα για το θέμα που μας απασχολεί. Αποδεικνύεται για μια, άλλη μια φορά ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στερείται ευελιξία. Όταν πρέπει να μεταφερθούν κάποιες πιστώσεις από ένα κονδύλι σε ένα άλλο για να ε, αντιμετωπιστούν προβλήματα επίγοντα ή απρόπτε. Το είδαμε, τι έγινε με την περίπτωση του ιού έμπολα. Χρειάστηκε πάρα πολύ ενέργεια και χρήμα για να μεταφερθούν οι πιστώσεις. Ε, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, την αποκατάσταση κτλ. Βάλανε χέρι σε εργαλεία όπως είναι η δημοσιονομική βοήθεια για την οικοδόμηση θεσμών στις χώρες, για να βοηθήσουν ε, τις χώρες αυτές. Ε, αλλά θέλω να τονίσω τελικά το εξής. όχι ως μέλος εδώ της Επιτροπής συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα ως βουλευτής και μέλος της σοσιαλιστικής ομάδας, ξέρω ότι το ζήτημα του προϋπολογισμού είναι ένα γενικότερο που κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε σοβαρά και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στις σχέσεις μας με το Συμβούλιο. Και να δούμε με ποιον τρόπο στο μέλλον θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε τέτοιες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με την απόκριση, αντιμετώπιση κρίσεων να έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα στην μεταφορά πιστώσεων από ό,τι είχαμε σήμερα. Um, Ευχαριστώ. Ο Σαρλ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω κάποιες απορίες, κυρίως για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο αλλά το ίδιο και για το γενικό προπολογισμό. Πρώτα απ' όλα για τη μείωση του προσωπικού. Εδώ και χρόνια ο ΣΑ και όχι μόνο ε, ε, ε, στα την προσοχή μας στο γεγονός ότι πρέπει η αναπτυξιακή πολιτική να είναι πρικοδοτημένη με έναν επαρκή αριθμό εργαζομένων για να υπάρχουν προγράμματα ποιότητας και αποτελέσματα ποιότητας. Δεν ξέρω κατά πόσον το έχουμε λάβει υπόψη αυτό διότι όταν γίνεται απολογισμό των φραγμών που προβάλλονται στον επαρκή αριθμό εργαζομένων δεν βρίσκονται η δικαιολόγηση είναι επαρκής. Και πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί στις ε, τριμερείς μορφές συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, δωρητή δικαιούχο μια χώρα αναπτυσσόμενη και μια τρίτη χώρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια παρέχει τεχνική βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζονται περισσότεροι εργαζόμενοι. Χρειάζονται πολλοί εργαζόμενοι, πολύ μεγαλύτερο προσωπικό για μια χώρα με την οποία έχουμε σχέσεις και δεδομένου ότι η αρχή της διαφοροποίησης θα πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της τρέχουσας περίοδου πρέπει να έχουμε έναν επαρκή ρυθμό εργαζομένων ιδίως για την τεχνική βοήθεια. Εμείς πάντοτε είχαμε τα σώμασταν υπέρ του να παίρνει στα χέρια τη σπιτάλη η τεχνική βοήθεια από την κλασική αναπτυξιακή βοήθεια. Και έπειτα για την ε, βοήθεια στον προπολογισμό. Αυτή είναι η δεύτερη μου παρατήρηση. Κατά τη δική μα ε, άποψη, αυτή η βοήθεια πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται σεβαστά κάποια κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια αυτά είναι η πρόθεση της κοινωνίας των πολιτών, η οποία πρέπει να ε, είναι διαρκής και η άλλη είναι η κοινοβουλευτική ανάπτυξη. Μπορεί η Επιτροπή σήμερα εν θερμό να μας απαντήσει σε, αυτό το, σε αυτή την ερώτηση ή έστω είναι διατεθειμένη να μας δώσει μια λεπτομερή περιγραφή της δημοσιονομικής στήριξης ε, προς την κοινωνία των πολιτών και την κοινοβουλευτική διάσταση στις δικαιούχους χώρες. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάουταλα και μετά τον κύριο Νόιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι είμαστε στο σημείο 7. Mm. Ωραία. 6 και 7 μαζί. Και οι δύο προπολογισμοί. Οι απαλλαγές. Τότε παρατηρήσεις και για τα δύο θέματα. Το θέμα του blending, της ανάμειξης, είναι για μένα ακόμη πολύ αμφιλεγόμενο, διότι όντως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια της παραχώρησης σε συνδυασμό με τα ιδιωτικά κεφάλαια, όμως ανησυχώ κάπως, διότι η Επιτροπή στηρίζει μόνο πολύ μεγάλης κλίμακας προγράμματα στην περίπτωση του blending, ιδίως για την ενέργεια. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε και να κοιτάξουμε επενδύσει να υπάρξουν και σε μικρής κλίμακας ε, αποκεντρωμένα και ε, διαδικτύωσης προγράμματα. Μόνο αυτά μπορούν να εκριζώσουν τη φτώχεια, ιδίω στι περιοχέ της υπαίθρου. Επίσης, οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου στην έκθεση του υπαριθμού 16 για το 2014 και για το blending αναφέρεται ότι οι ενδείξεις ότι έγιναν επενδύσεις χωρίς συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μάλλον μια σοβαρή παρατήρηση. Σημαίνει ότι τα κονδύλια της παραχώρησης δεν είναι απαραίτητα σε αυτή την περίπτωση. Και στην περίπτωση του blending μας απασχολεί πολύ κατά πόσον είναι αποτελεσματικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και όπως λέει το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να δούμε τον ε, μηχανισμό ε, των κονδυλίων ε, για το blending σε συνδυασμό με την αιρεσιμότητα Νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και ότι το ευρωπαϊκό blending δεν μπορεί να αρκεί μόνο του για την ε, αποτίμηση των ε, των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών προγραμμάτων στα πλαίσια τη επίσημης αναπτυξιακή βοήθεια. Όπω είπε και ο κ. Γκέρεν, υπάρχει μια νέα συμφωνία για τη δημοσιονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Επίτροπος Πίμπαλξ μίλησε για συμβάσεις καλής διακυβέρνησης. Κάτι που προσαγγίζει πολύ αυτό που είπε ο κύριος Γκέρενς. Η βοήθεια στον προπολογισμό θα πρέπει να υπόκειται σε κριτήριο ανάπτυξη τη κοινωνία των πολιτών, μεγαλύτερη συμμετοχή τη και τη κοινοβουλευτική διάσταση. Διότι και στι δύο περιπτώσει ο ρόλο του είναι πολύ σημαντικό ω προ τη λογοδοσία λογοδοσία που καμιά φορά είναι και το μεγαλύτερο θέμα ε, ως προς την στήριξη του προπολογισμού. Αυτές τις παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Ευχαριστούμε κύριο Νόιζερ. Ε, ich möchte nur ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen, weil ich denke, dass... Ε, μια παρατήρηση θέλω να κάνω και κάποια σχόλια. Καλή είναι η συζήτηση που κάνουμε, αλλά υπάρχει διαρκής υποχρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας τα κράτη-μέλη έχουν μειώσει την αναπτυξιακή τους βοήθεια στον προϋπολογισμό τους και αυτό έχει επίδραση και στη δική μας πολιτική. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα κράτη-μέλη μας. Αν δούμε τις στατιστικές της Eurostat και τις πιστέψουμε, τις πιστεύω, 80% του πληθυσμού στην Ευρώπη είναι υπέρ της καλής αναπτυξιακής πολιτικής που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μας για το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αρχής και θα πρέπει πάντα να το τονίζουμε και να το θέτουμε υπόψη και στα κράτη-μέλη και να αγωνιζόμαστε να μας δίνουν ε, τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Για την στήριξη του προπολογισμού ε, έχει σημασία στις αναψώμενες χώρες οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρα πολύ συγκεκριμένα και με ακρίβεια να ελέγχουν αν λειτουργεί η μακροοικονομική βοήθεια τα χρήματα που δίνουμε για την ενίσχυση του προπολογισμού. Εκεί θα πρέπει να έχουμε στοιχεία αξιόπιστα και εκεί θα πρέπει να κάνουν τους ελέγχους οι αντιπροσωπείες της Ένωσης επιτόπου. Ε, το επόμενο. Ακούω ε, βέβαια ε, με μισόλογα από τις αντιπροσωπείες εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το τι σημαίνουν οι περικοπές επιτόπου. κόβονται προγράμματα ε, αποδυναμώνονται, αφεμάσονται προγράμματα, παρακαλούνται οι ΜΚΟ να μεταθέσουν τα προγράμματά τους για το επόμενο έτος, παρακαλούνται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να κάνουν προκαταβολές οι ίδιες. Είναι μια κατάσταση που είναι τελείως αφόρητη και καθόλου ικανοποιητική για την πρακτική δουλειά επιτόπου. Δυστυχώς, κανένας από τους αντιπροσώπους ε, εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βγαίνουν να τα πούν αυτά δημόσια. Ε, στα λένε με μισόλογα και ψιθυριστά ε, όταν πας ως βουλευτής σε ταξίδια αποστολές. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια αντιμετώπιση τόσο φιδωλή, για να μην πω ε, τόσο τσιγκούνικη αντιμετώπιση. Ε, χρειάζεται να συνεχίζουν τα προγράμματα με την ίδια ένταση και τους ίδιους ρυθμούς που είχαν στο παρελθόν. Αυτά θα πρέπει να τα πούμε στη γενικότερη συζήτηση για τον προπολογισμό. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ο Ερίκη και πάλι. Μία ερώτηση επιπλέον έχω. Το ελεγκτικό συνέδριο επισημαίνει ότι τα σφάλματα ή η κακή διαχείριση κάποιες ατασταλίες στα προγράμματα είναι της τάξης ε, του 3,5%. Το ποσοστό αυτού του σφάλματος δεν είναι τραγικό. Βέβαια, δεν είναι και ασήμαντο. Και σίγουρα δεν υπάρχει βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες χρόνιες. Κανονικά, μετά από τις προειδοποίησεις ε, και τις επισημάνσεις που κάνει το ελεκτικό συνέδριο για κακή διαχείριση σφάλματα, θα πρέπει να βελτιώνεται το ποσοστό σφάλματος. και έστω και σταδιακά να υπάρχει μια βελτίωση, μια μείωση του ποσοστού σφάλματος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μεριμνήσει ότι στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις που κάνει των διαφόρων σχεδίων και προγραμμάτων να μην δέχεται τόσο υψηλά ποσοστά σφάλματος η ε, κακής διαχείρισης, δηλαδή του ύψους 3,4%. Μάλιστα. Πληθώρα ερωτήσεων. Καταρχήν, ερώτηση Γκέρνς ε, για την ε, έλλειψη προσωπικού και ε, τον αντίκτυπο στις διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, δημοσιονομική στήριξη, ρώτησε ο κύριος Νόιζερ, και πώς επηρεάζει την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού ή πώς ενισχύει την κοινωνία των πολιτών. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Τον Ιανουάριο θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΦΚΟ για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τη δημοσιονομική στήριξη. Οπότε μπορείτε να του παραπέμψετε αυτά τα ερωτήματα. Συγκεκριμένη ερώτηση για το blending, το συνδυασμό δανείων επιχορηγήσεων. Επίσης, για το που κάποιες επιλογές πολιτικής, που θα πρέπει να αφιερώνουν τα κονδύλια είναι θέμα όχι τόσο ελέγχου όσο επιλογής πολιτικής για ενεργειακά προγράμματα. Επίσης, πώς συνδυάζεται ο συνδυασμός αυτός στο blending με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, το ODA. Και τι εμπίπτει στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και τι όχι. Φαντάζομαι θα τα σχολιάσει αυτή. Επίσης, το θέμα της υποχρηματοδότησης, των δημοσιονομικών προβλημάτων, της ε, έλλειψης ε, κονδυλίων, της αναντιστοιχίας ε, δεσμεύσεων ε, ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών, της ε, έλλειψης πιστώσεων πληρωμών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχετικά υψηλό ποσοστό σφάλματος και αν μπορούμε να το βελτιώσουμε, να το μειώσουμε. Ο κύριος Λαγκού από την ε, Μπαγκού, μάλλον, από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Επειδή πρώτη φορά σε βλέπουμε στην Επιτροπή, πείτε μας δύο λόγια για το ποιος είστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ονομάζομαι Λίκ Μπαγκούρ. Είμαι διευθυντή σε θέματα πόρων στην Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Σας ευχαριστώ για τη σχετικά θετική σας γνωμοδότηση για τη διαχείριση των αναπτυξιακών πολιτικών, είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου, είτε μέσω του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας στα πλαίσια του Γενικού Προϋπολογισμού. Το ποσοστό του σφάλματος είναι σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων και λαμβάνουμε υπόψη μετά από εξονυχιστική ανάλυση της παρατηρήσης του ελεκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να δείξουμε βέβαια ότι η αρρωγή που παρέχουμε ευθυγραμμίζεται με τους πολιτικούς μας στόχους. Είναι πολύ σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά τη σωστή χρήση των κονδυλίων. Δηλαδή όχι, θα, δεν θα πρέπει μόνο να έχουμε χρηστή και σωστή διαχείριση, αλλά και αυτά αποτελέσματα. Εξού και η επίκαιρη σημερινή συζήτηση για την αποτελεσματικότητα τη αναπτυξιακή μα βοήθεια. Επανέρχομαι στη διαχείριση. Το ποσοστό σφάλματο είναι 3,4%. Ε, μία μικρή αύξηση. Αλλά γενικά μειώνεται. Στο συνολικό προπολογισμό είναι κάτω από το 3%. Πολύ θετικό μήνυμα. Είχαμε διαφωνία για δύο σφάλματα με το ελεκτικό συνέδριο και αυτό επηρέασε ε, αυτό το ποσοστό Αλλιώ αν δεν είχαμε αυτές τι δύο διαφωνίε, είχαμε σαφώ χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος. Και μάλιστα στην Επιτροπή Ελέγχου προπολογισμού, καταθέσαμε όλα τα επιχειρήματα από πλευράς ΕΚΟ. Θεωρούμε πάντως ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αποδεικνύει ότι το γενικό σύστημα ελέγχου είναι καλό στη θεωρία. Η έμπρακτη εφαρμογή του θα πρέπει κάπως να βελτιωθεί. Ε, αυτό επιβεβαίωσε και η δική μας μελέτη για το εναπομείναν ποσοστό σφάλματος. Όπως επισημαίνετε και εσείς στην γνωμοδότησή σας, κυρία Πρόεδρε, μερικά σφάλματα αφορούν διεθνείς οργανισμούς. Είτε γιατί δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για τη χρήση των κονδυλίων, είτε γιατί δεν παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για τις διάφορες δραστηριότητες. Επίσης έχουμε προβλήματα με κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είναι δικαιούχοι επιχορηγήσεων και δεν σέβονται πάντα όλους τους όρους των συμβολέων. Πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε και μεριμνούμε ώστε να αναβελτιώσουμε την διαχείριση των κονδυλίων, ιδιαίτερα μετά το πρόγραμμα δράσης του 2013 και την αιτήσια έκθεση δραστηριοτήτων που έχει υποβάλει ο διευθυντής της ΔΕΦΚΟ. Τώρα για τη δημοσιονομική στήριξη. Ο κύριος Δεμέλο θα έρθει, ο Γενικός Διευθυντής, στην Επιτροπή σας τον Ιανουάριο για να σας ενημερώσει ειδικά για το θέμα αυτό. Οπότε δεν θα είμαι εδώ εξαντλητικός. Πάντως για 55 ε, συναλλαγές ε, ε, που εξέτασε το ελεκτικό συνέδριο, τρία σφάλματα μόνο εντοπίστηκαν, ενώ πριν από τρία χρόνια είχαμε 20. Υπάρχει αισθητή βελτίωση στη δημοσιονομική στήριξη, χάρη στη μεταρρύθμιση του 2011 που έκανε η ΔΕΦΚΟ σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Όντως, είναι υποχρηματοδοτούμενη η αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτό από τα τέλη του 2013. Στα τέλη του 2014, σε ό,τι αφορά τη γενική μας διεύθυνση, την ΤΕΦΚΟ, μεταφέραμε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ απλήρωτους λογαριασμούς στην επόμενη χρονιά, το 2015. Οπότε, πέρασαν αυτά εκτός της πολιτικής γειτονίας στην διεύρυνση, στην Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης και χρησιμοποίησαμε το μέσο ευελιξίας ε, για να κάνουμε όσο, πιο μεταφορές, όσο περισσότερες μεταφορές μπορούμε μεταξύ των δημοσιονομικών γραμμών και των κεφαλαίων για να καλύψουμε τις ανάγκες. Και μάλιστα κάναμε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και χρηματοδοτήσαμε τα πιο σημαντικά προγράμματα κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους πιο ευπαθείς εταίρους μας. Η μεταφορά βέβαια 700 εκατομμυρίων στον επόμενο προϋπολογισμό και ο προϋπολογισμός για το 2015 ε, δεν μπορεί και πάλι να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της αναπτυξιακής πολιτικής. Τώρα, μείωση του προσωπικού. Ισχύει, είναι κάτι που είχαμε προβλέψει εδώ και πολύ καιρό 2% μείωση το χρόνο των υπαλλήλων μας και 1% στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 1% για τις ε, εσωτερικές ανακατατάξεις. Για τη γενική διεύθυνσή μας, με εξαίρεση την πολιτική γειτονία, είναι 22 λιγότερες θέσεις για το 2015 και το ίδιο για το 2016 και το 2017. Κάθε χρόνο θα χάνουμε 22 θέσεις, μόνο για τους υπαλλήλους, τους μονίμους. Τώρα, τα περισσότερα κονδύλια για τις δραστηριότητες έχουν μπλοκαριστεί στα επίπεδα τα ονομαστικά του 2005, οπότε περιορίζουμε και τους συμβασίουχους. Ε, έχουμε 7 λιγότερους συμβασίουχους κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά ως προς τη μείωση του προσωπικού. Αλλά αυτή η μείωση του προσωπικού μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασιών μας. Γι' αυτό και λάβαμε κάποια μέτρα για τη προηγούμενη μελέτη του επιμερισμού του φόρτου εργασιών ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπάλληλοι στις, στα σχέδια προτεραιότητας και στις ώρες προτεραιότητας. Για παράδειγμα, δώσαμε έμφαση στις χώρες της γειτονίας και στην Υποσαχάριο Αφρική και όχι τόσο στη Λατινική Αμερική. Επίσης, έχουμε μόνιμη παρακολούθηση του προσωπικού των αντιπροσωπιών εφαρμόζουμε το σύστημα Optimus και κάθε χρόνο με βάση την περιτροπή, την περιτροπής χρήση των υπαλλήλων μπορούμε να ε, συγκεντρώνουμε το προσωπικό στις προτεραιότητές μας. Έχουμε όντως έλλειψη προσωπικού, αλλά προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το προσωπικό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα για το blending, το συνδυασμό των μέσων, συνδυασμό δανείων επιχορηγήσεων ξεκίνησε με τη γειτονία με τη διευκόλυνση της γειτονίας, μετά προβλέψαμε αντίστοιχους μηχανισμούς και σε άλλες γεωγραφικές ζώνες, κατά τα τέλη του προηγούμενου Πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε μία αύξηση της σημασίας του blending. Βέβαια, σε σχέση με τα κονδύλια της αναπτυξιακής ε, βοήθειας δεν είναι τόσο σημαντικό το επίπεδο του blending. Αλλά είναι σημαντική η μόχλευση του blending και κυρίως ε, κινητοποιούμε κάποια κονδύλια πέραν των πιστώσεων. 1 προς 15 είναι η μόχλευση του blending, μερικές φορές και 1 προς 20. Για ένα ευρώ που επενδύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στο συνδυασμό των μέσων, ε, ανακτούμε 20 ευρώ. Και μπορούμε να βρούμε και επιπλέον χρηματοδότηση. Και είμαστε ευγνώμονες προς το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεση με θέμα το blending και φυσικά θα αναλύσουμε διεξοδικά τα πορίσματα και τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου και θα τις λάβουμε υπόψη προκειμένου να αναλύσουμε περιπτωσιολογικά την προστιθέμενη αξία του συνδυασμού των μέσων, του blending, προκειμένου να αποφύγουμε επικάλυψη η κεροσκοπία και τα μέσα του blending πραγματικά να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που χωρίς επιχορηγήσεις δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν διαφορετικά. Αυτά και νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Um, Τώρα το σκέφτηκα, είπατε ότι θα διαβιβάσετε αυτή την πληροφόρηση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σε εκείνους απαντήσατε, είπατε, γιατί σας ρωτάνε για τα έργα, τα διάφορα, τα project. Μήπως θα μπορούσατε να στείλετε και σε εμά ε, μια ενημέρωση. Βάλτε μας ε, ένα αντίγραφο και εμάς, δεν γίνεται. Γιατί θα συμπροεδρεύσω εγώ την Πέμπτη για την IT θα είμαι παρούσα και έχει σημασία και τα δικά μας μέλη να ενημερωθούν σχετικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ε, σήμερα μπορούμε να σας στείλουμε τις απαντήσεις που στείλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου. Ευχαριστώ. Κοντ, Κοκομπού, κάθε, μέρα, κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν όνομα. Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού λοιπόν έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της δεν λέγεται πια κόκομπι. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο, δεν βλέπω κανέναν για αυτό το σημείο. Προθεσμία κατάθεση τροπολογίων, Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε 21 Ιανουαρίου. Σας παρακαλώ, ελάτε την Πέμπτη το πρωί, αν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, θα είναι και η Επιτροπή και θα ε, εξηγήσει πλήρω ορισμένε από τι απαντήσει αυτέ και θα ψηφίσουμε 21 του μηνό Ιανουαρίου του 2015. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 8 που είναι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και η συγκήτριά μας είναι η κυρία Χάιντι Χάουταλα. Είναι καθιστική ε, πρακτική ε, μαζί με την έκθεση Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να δίνουμε και εμείς μια ε, έκθεση. Ε, εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις 23 Ιουνίου του 2014 αυτό και αφορά το έτος 2013. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς να πούμε τη γνώμη μας για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει παγκοσμίως ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, θα δώσω μέσα στο λόγο στην κυρία Χάουταλα, τη συντάκτη της γνωμοδότησης, για να μας την παρουσιάσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνέταξα την έκθεση αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και γι' αυτό το σχέδιο απεστάλλει στις μεταφραστικές υπηρεσίες και προέκυψαν λίγες αλλαγές εντωμεταξύ στο σχέδιο της έκθεσης. Θα έχει συμβεί και σε άλλες εκθέσεις αυτό, αλλά να εξηγήσω λίγο αυτές τις επιπλέον αλλαγές στη συνέχεια μετά. Είναι πολύ σημαντικό η έκθεση για την οποία είναι υπεύθυνο ο κ. Παντζέρη στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι σημαντικό να αναφέρει τις ε, παρατηρήσεις μας για την ευρωπαϊκή πολιτική για την για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε συζητήσεις μεταξύ μας και βλέπω ότι και η δική του συλλογιστική θέλει να καλύπτει την ε, αναπτυξιακή πολιτική στην κυρίως έκθεση, την δική του, που συντάσσεται στην, υπό την αιγύδα της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Να επαναλάβω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η παρατήρηση είναι υψή τη σημασίας. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναπτυξιακή της συνεργασία τη βασίζει στην προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία πρέπει να υλοποιείται. Να ευαισθήσω εδώ την προσοχή στο ρόλο των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες εταίρους. Και όλων γενικώ των παγκοσμίων οργανισμών που μπορεί να είναι δωρητέ και εταίροι. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δουν ακριβώς την αναπτυξιακή βοήθεια υπό τη σκοπιά της προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θεματολόγιο για μετά το 2015, όπου ήδη έχει τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο, πρέπει επίσης να αναφερθεί, καθώς τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εξορθολογιστούν στο πλαίσιο του ε, διαστήματος μετά το 2015, με νέους ε, συγκεκριμένους στόχους υπό τον κατάλογο των ε, αναπτυξιακών στόχων τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα πρέπει και πολιτιστικά μάλλον δικαιώματα πρέπει να καλύπτονται και θα πρέπει να τους δώσει κεντρική διάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωτερικέ της σχέσεις, προωθώντας και τα εργασιακά δικαιώματα και πρότυπα, τη σχετικά νέα προσέγγιση για τα κοινωνικά δικαιώματα και για την εκρίζωση της πτώχειας και να υπάρχουν λειτουργικέ κοινωνικέ ρήτρε σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τέτοιε, αλλά δεν είναι πάντοτε δεσμευτικέ. Επίση ήθελε να υπάρχει ένα εδάφιο για τι εταιρείε και το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ υποστηρίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νομικό δεσμευτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συγκεκριμένη ανάγκη να αναζητήσουμε τα ανάλογα ένδικα μέσα, ώστε εφόσον υπάρχουν σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προβλέπονται και ανάλογε κυρώσει και η δυνατότητα προσφυγή των θυμάτων τέτοιων παραβιάσεων. Αυτέ είναι κάποιε προκλήσει λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνέ δίκαιο. Έπειτα έμφαση δίνω και στην ε, πολιτική συνεργασία για την ανάπτυξη. Η νέα είπατε εκπρόσωπος, κυρία Μαγκερίνη, έχει την αρμοδιότητα και ενδιαφέρεται να προωθήσει τους πολιτικούς στόχους για την ανάπτυξη και θα πρέπει να τις θυμίζουμε ότι αυτό είναι και για μας ε, ένα κύριο μέλημα των εξωτερικών μας, θα πρέπει να είναι ένα κύριο μέλημα των εξωτερικών μας σχέσεων και της πολιτικής τους. Ένα παράδειγμα για το εμπόριο είναι ότι όταν έχουμε πρωτισμισιακές ευρωπαϊκές συμφωνίες όπως το GSP+, θα πρέπει να έχουμε και τους ανάλογους μηχανισμούς υλοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφόσον μπορεί να υπάρξουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά για τη χρήση της γης και για τα σχετικά δικαιώματα. Νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα εδώ, διότι συνδυάζουμε πάλι την ανάπτυξη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτείνω να αναζητήσουμε δεσμευτικές κατευθυντήρες δαμές για να αποφύγουμε την αρπαγή γεών. Και θα πρέπει να ε, γίνει και η παραπομπή στις συστάσεις του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για το δικαίωμα στα τρόφιμα με μια σημαντική μετατόπιση της ε, ε, οικολογικής προσέγγισης στη γεωργία ως ένα μέσο διατήρησης του δικαιώματος του επισητισμού. Και να μην ξεχνάμε και τη σχετική έκθεση για τον υποσιτισμό. Αυτό το θέμα πρέπει να το έχουμε υπόψη και το λέω σε όλους σας. Η υποβάθμιση στη χρήση της γης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εάν δεν το έχουμε κατά νου και δεν έχουμε και μια οικολογική προσέγγιση στην παραγωγή τροφίμων, θα υπάρξουν ε, πολλές σπατάλες και πολλά θα πάνε χαμένα. Έπειτα και η ανάπτυξη της ασφάλειας πρέπει να συνδυαστεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ευαίσθητες και να δίνουν προσοχή στα στις πρώτες ενδείξεις για σοβαρές σειράξεις οι συγκρούσει που μπορεί να έχουν σοβαρότατε επιπτώσεις για την ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο της ασφάλεια τη ανάπτυξη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτείνω να αναφέρουμε τις πλέον ευάλωτες ομάδες που θα πρέπει να προστατεύονται. Δηλαδή γυναίκες, άνθρωποι με αναπηρίε και παιδιά θα πρέπει να χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή στι προσπάθειε ανακούφιση αποκατάσταση και ανοικοδόμηση. Τέλος, υπάρχει ένα εδάφιο για την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να βεβαιωθούν ότι ο νόμος ε, για το άσυλο, τον έλεγχο των συνόρων πρέπει να γίνονται σεβαστά και μια ιδιαίτερη μνήα γίνεται και για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ε, φυσικών πόρων. Και εδώ τα δικαιώματα των αυτοχθονών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στην Βερμανία Μιανμάρ λόγου χάρη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους αυτόχθονες και τη χρήση της γης σε περιοχές όπου οι πολυεθνικές ετοιμάζονται να κάνουν επενδύσεις και να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους τους φυσικούς πόρους της χώρας. Και μετά υπάρχουν και μερικές αλλαγές στην επόμενη εκδοχή της έκθεσης, κυρίως διατύπωσης για το τμήμα που αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την άδειά σα, θα πρότεινα να στηρίξουμε την ιδέα οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ορυκτά των συγκρούσεων να λάβουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ιδάλλως, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του. Λόγω χάρη αυτά που συμβαίνουν στο Ανατολικό Κονγκό και τον πόλεμο που μένεται εκεί. Αυτά λίγο πολύ είχα να σας προτείνω. Σε... σας ευχαριστούμε. Όντω η νέα είπατε εκπρόσωπος η κυρία Μαγκερίνη έχει συμφωνήσει να έρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην Επιτροπή μας. Οπότε θα θέσουμε και τα θέματα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ό,τι άλλο χρειαστεί. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουμε κάποια ημερομηνία, αλλά έχουμε χρόνο, θα το προβλέψουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ καλά τα νέα. Να δούμε ποιο θέλει το λόγο, οι σκιώδεις εισηγητές. Δεν ξέρω αν είναι όλοι εδώ. Η Μαρίνα Αλμπιόλ Γκούσμαν τη Γκου έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δείξουμε τι σημασία έχει η συνεργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να πούμε ότι μισή σελίδα μόνο αφιερώνει ε, η έκθεση για τη θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό είναι αξιοσημείωτο από μόνο του. Επίση, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το βασικό εμπόδιο για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάπτυξη στι χώρε αυτέ είναι οι συμφωνίες που του επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρε που φτωχοποιούνται, επιβάλλουν το ελεύθερο εμπόριο, δεν λαμβάνουν υπόψη του τι οικονομικέ ασυμμετρίε, σαφεί και συγκεχημένε αναφορέ και όχι δεσμευτικέ μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, χρησιμοποιούν ως εργαλείο, ως ένα ακόμα εργαλείο ε, αυτές τις συμφωνίες για εμπορικές συμφωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ε, πέφτουν στο βωμό οικονομικών συμφερόντων που αφιερώνεται άπειρος χρόνος και ενέργεια και χρήματα εκεί και δίνουν σε ε, εκατομμυριούχους ε, πολυεθνικές τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται όχι μόνο τους φυσικούς πόρους αλλά και τους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα τονίσουμε. Μα τι μιλάμε για σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόθεση τους ενώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί η αναπτυξιακή βοήθεια ως μέσο εκβιασμού των φτωχοποιημένων χωρών να αναγκαστούν να δεχθούν ε, ε, συμφωνίες που κάνουν τη χώρα τους ξέφραγο αμπέλη για τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές ατιμωρησίες στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, απουσία εργατικών δικαιωμάτων, ε, καταπίεση. Αυτά κάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές πολυεθνικές στις χώρες που έχουν φτωχοποιήσει οι ίδιες. Και τελικά φυσικά δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την ε, πολιτική οδό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που θα κάνει είναι να αναγκάσει τις χώρες να δεχτούν αυτές τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Εμείς θεωρούμε ότι αν θέλουμε πραγματικά η πολιτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να είναι εγγυημένα τα ανθρώπινα δικαιώματα στις φτωχοποιημένες χώρες θα πρέπει εμείς να τις βοηθήσουμε από την Επιτροπή μας εδώ για τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εν λόγω χώρες. Ας πούμε να αρχίσουμε από την ε, συμπεριλήψη ε, δεσμευτικών ρητρών